Madame Κύριε Κραπίνη, κάτι θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Βέλγο Πρωθυπουργό, ε, κάποιος συνάδελφος είπε το εξής. είπε ότι οι γυναίκες δεν γράφουν την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ναι, φυσικά ε, δεν ήταν σωστό αυτό που υπόθηκε. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω